Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και το Ουγγρικό Δικαστήριο ανέστηλε τη αγωγή κατά την κυρία Τζόμπαν γιατί αποσύρθηκε αυτή, αυτό το αίτημα και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή, το αίτημα άρσης ασύλη